Ladies and gentlemen, please. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ καθίστε, έχει θέσεις πίσω. Good morning. Καλημέρα σας και καλωσορίσατε στην κοινή αυτή συνεδρίαση της Επιτροπής μας και της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Θα αρχίσω εγώ ως πρόεδρος της Υποεπιτροπής, αλλά θέλω να καλωσορίσω και τον πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών, Διουσόν και θα κάνουμε μία πρώτη ανταλλαγή απόψεων για τη χρηματοδότηση της ΚΠΑΣΑ. Έχουμε εισηγητές και των δύο επιτροπών εκ μέρους της δικής μας τον κύριο Κούκαν και εκ μέρους της Επιτροπής Προϋπολογισμών τον κύριο Ιντρακτοράν. Επίσης έχουμε έναν εξέχοντα εμπειρογνώμονα Βαρβιάν Περπέν που θα μας μιλήσει ήδη από την αρχή αλλά πρώτα θα δώσω το λόγο στον πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών κύριο Ζαν Αρτουή. Madame la Présidente, Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι ιδιαίτερα για την κοινή μας αυτή αποστολή. Στην Επιτροπή Προϋπολογισμών θέλουμε να συμβάλλουμε και εμείς στην αποτίμηση, στην εκτίμηση της ευρωπαϊκής πολιτικής ασφαλείας και άμυνας. και θα θέλαμε χάρη στις δεδομένα που αφορούν τον προϋπολογισμό να εκποτιμήσουμε το εύρος των δραστηριοτήτων που αναλαμβάνονται και τα περιθώρια που έχουμε αλλαγής προόδου και ελιγμών για να μπορέσει η Ευρώπη, για να δούμε αν η Ευρώπη μπορεί να αναλάβει όλα όσα έχει υποσχεθεί σε θέματα ασφαλείας και άμυνας. θα ήθελα να σας ε, παρουσιάσω τον ε, προσκεκλημένο μας. ο οποίος ε, δραστηριοποιείται στο Ινστιτούτο για Πολιτικές Επιστήμες στη Γκρενόμπλ και είναι και επισκέπτης καθηγητής στην Πολωνία, στο Ευρωπαϊκό Κολέγιο. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτέ. Με μεγάλη χαρά θα σας κάνω την παρουσίασή μου σήμερα για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και αποστολών της ΚΠΑΣΑ. Σε τρία μέρη θα κάνω την παρουσίασή μου. Πρώτον, τι χρηματοδότηση υπάρχει. Δεύτερον, ποια προβλήματα παρατηρούνται. Και τρίτον, η προοπτική μελλοντικών εξελίξεων. Για την υπάρχουσα την τωρινή χρηματοδότηση είναι κατακαιρματισμένη και πολύπλοκη νομίζω διότι υπάρχει ο διαχωρισμός μεταξύ πολιτικών αποστολών, μη στρατιωτικών δηλαδή, που, αφορούν, που προέρχονται από τον ενωσιακό προϋπολογισμό, αλλά μπορούν να χρηματοδοτηθούν και από ατομικές εισφορές των χωρών μελών, όπως αποφασίσει το Συμβούλιο, και από την άλλη τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται κυρίως από τα κράτη-μέλη με μονομένο ατομικό τρόπο με βάση την αρχή costs lie where they fall. Υπάρχει και χρηματοδότηση από τον μηχανισμό της Αθηνάς. Δηλαδή με βάση χρηματοδότηση ορισμένων τμήματων του κόστους από την Αθηνά. Ο μηχανισμός αυτός, σας υπενθυμίζω, είναι μηχανισμός που περιορίζεται στη χρηματοδότηση τμήματος του κοινού κόστους από τα κράτη-μέλη αλλά με βάση μία κλίδα κατανομής ανάλογα με το ΑΕΠΤΟΝ και σε πλαίσιο που παραμένει διακυβερνητικό. Η Αθηνά είναι διακυβερνητικό δηλαδή όργανο και εργαλείο χρηματοδοτεί ένα μικρό τμήμα του κόστους των επιχειρήσεων, 10 με 15% και ορισμένο τμήμα του κόστους αυτού υποχρεωτικά χρηματοδοτείται από την Αθηνά, ενώ το υπόλοιπο χρηματοδοτείται μόνο αν η Ειδική Επιτροπή της Αθηνάς ή το Συμβούλιο το αποφασίσει. Τι προβλήματα μπορούν να ταυτιστούν εδώ με βάση αυτό τον πολύπλοκο μηχανισμό χρηματοδότησης. Τρία πρώτον θέμα αποτελεσματικότητας ή μάλλον έλλειψης αυτής. Θέμα δημοκρατικού ελλείμματος και τρίτον η λογική της αλληλεγγύης, η έλλειψης αυτής. Πρώτα λοιπόν η έλλειψη αυτης ή μάλλον η αναποτελεσματικότητα. Καταρχήν οι πόροι που διατίθενται για τις αποστολές και επιχειρήσεις είναι περιορισμένη στον ευρωπαϊκό και στους εθνικούς προϋπολογισμούς υπάρχουν περιορισμοί. Γενικά λοιπόν όταν αναλαμβάνεται, αποφασίζεται μία επιχείρηση πάντα υπάρχουν προβλήματα για την χορήγηση διάθεση των πόρων. Τα κράτη διστάζουν πάρα πολύ να συμβάλλουν και η δημιουργία των δυνάμεων για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις είναι επίσης δύσκολη. Σας υπενθυμίζω ότι η Αθηνά χρηματοδοτεί μικρό τμήμα το κόστος αυτού, διότι και αυτή έχει πολύ περιορισμένους πόρους. Δεύτερο πρόβλημα. πάντα για την Η ταχύτητα της ανάδρασης ή αντίδρασης. Ε, η ταχύτητα του μηχανισμού λήψης αποφάσεων είναι πολύ μικρή, χαμηλή και για τις πολιτικές και για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις για λόγους που οφείλονται στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και παρά τους μηχανισμούς που υπάρχουν για μια άμεση χρηματοδότηση των πολιτικών τουλάχιστον επιχειρήσεων ή για τις στρατιωτικές για την προχρηματοδότηση που θα επέτρεπε μια πιο γρήγορη διάθεση πόρων στα πλαίσια της Αθηνάς με μορφή όμως προχρηματοδότησης και μόνο από την Αθηνά. Δεν μιλάω για τις εισφορές εκτός Αθηνάς. Άλλο πρόβλημα επίσης πάλι αναποτελεσματικότητος η εξωτερική συνοχή. Το κατακαιρματισμό των τρόπων και πολλαπλασιασμό των τρόπων χρηματοδότησης δεν συμβαδίζει και πάρα πολύ με την ιδέα κάποιας εξωτερικής συνοχής ή συνέπειας και αυτό παρόλα αυτά επαναλαμβάνεται πολλές φορές στη συνθήκη ως όρος, αλλά δεν συμβαδίζει με την πολιτική λογική της σφαιρικότερης αντιμετώπισης που ζητούν πολλά κείμενα. Από τη μια δηλαδή κατακαιρματισμό των πόρων και από την άλλη απέτηση συνοχής και ολοκληρωμένης προσέγγισης. Αυτά δεν συμβαδίζουν νομίζω. Άλλο πρόβλημα, <clears throat> δεύτερο είδος προβλήματος, όχι πια η αναποτελεσματικότητα, αλλά η ανεπάρκεια δημοκρατικών εγγυήσεων. Οι πολιτικές επιχειρήσεις ελέγχονται πολιτικά και άρα έτσι ανταποκρίνονται σε αυτό το κριτήριο. Καμιά φορά σημειώνονται δυσκολίες ως προς τη διαφάνεια των επιχειρήσεων αυτών γιατί η εγγραφή αυτών των επιχειρήσεων στον προϋπολογισμό δεν γίνεται πάντοτε με τον διαφανέστερο δυνατό τρόπο. Και επίσης και κυρίως υπάρχει το πρόβλημα της έλλειψης ελέγχου, κοινοβουλευτικού ελέγχου για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και του μηχανισμού της Αθηνάς. Εκτός αυτού, ο μηχανισμός αυτός ή μάλλον η πληροφόρηση που χορηγείται στο Κοινοβούλιο για την Αθηνά εξαρτάται αποκλειστικά από το Συμβούλιο. Τρίτο είδος προβλήματος, κατηγορία προβλημάτων, εσωτερικό πρόβλημα αλληλεγγύης. Δεν υπάρχει, δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχουν τα κράτη-μέλη στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και εδώ τίθεται το πρόβλημα της αλληλεγγύης. Τα κράτη-μέλη γενικά είναι λίγα τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν τακτικά σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Και όσο περισσότερο φορές συμμετέχει ένα κράτος σε μια επιχείρηση, σε, επιχειρήσεις, τόσο περισσότερο κόστος αναλαμβάνει βέβαια. Εξού και η έκκληση των πιο δραστηρίων χωρών που συμμετέχουν για καλύτερη κατανομή του άχθους. Και απ' την άλλη, τα κράτη που συμμετέχουν θεωρούν τα μη συμμετέχοντα κράτη κατά κάποιον τρόπο σαν free riders. Δηλαδή, κράτη που δεν αναλαμβάνουν δίκαια ή ισότιμα το πολιτικό και οικονομικό ρίσκο ενώ θα επωφεληθούν ίσως από τα αποτελέσματα. Έρχομαι τώρα στο θέμα των πιθανών εξελίξεων για το μέλλον και αυτές σε τέσσερα σενάρια τις έχω μοιράσει. Πρώτον, αυτό που μπορούμε να συζητήσουμε πιο σύντομα την υπόθεση ότι δεν αλλάζει τίποτε, Στάτους κουβό. Αυτό το σενάριο είναι πιθανό. Αν θέλουμε να βελτιωθεί η επιχειρησιακή δυνατότητα της ε, ΚΠΑΣΑ, τότε φυσικά δεν πρέπει να παραμείνουμε στο status κουβό. Αλλά βέβαια, ε, όπως γνωστόν, υπάρχουν προβλήματα που το καθιστούν πιθανό αυτό το σενάριο. Τι άλλες υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε. Ας πούμε, να συγκεντρωθούν περισσότεροι μηχανισμοί στα πλαίσια ενός ταμείου εκτός προϋπολογισμού. Δηλαδή να μεταφερθούν θέσεις του προϋπολογισμού από τον ενωσιακό προϋπολογισμό προς την Αθηνά έτσι ώστε τα μεμονωμένα κρατικά κόστη να περάσουν στην Αθηνά. Αυτό δεν είναι πολύ ρεαλιστικό, γιατί η έξοδος από τον προϋπολογισμό δεν μου φαίνεται ρεαλιστική. όλα αυτά, παρόλα αυτά, αλλά βλέπουμε ότι τα κράτη-μέλη, μερικά από αυτά, μπορεί να έχουν αυτό το πειρασμό μεταφοράς ορισμένων δαπανών από τον προβλογισμό προς την Αθηνά. Και άρα το σενάριο αυτό, αν και δεν είναι επίσημο στόχος κανενός, παραμένει πιθανό, δυνατό. Τώρα τα υπέρ και τα κατά. Λίγα είναι τα υπέρ, πολλά τα κατά. μπορεί να υπάρξει κίνδυνος ασυνέπειας, δηλαδή πολλές δαπάνες για την ΚΠΑΣΑ πρέπει να συνδεθούν και με τις γενικότερες δαπάνες εξωτερικής πολιτικής που δεν ανήκουν στην ΚΠΑΣΑ και ιδίως πρόβλημα δημοκρατικού ελέγχου και αποτελεσματικότητας. Άρα και αυτό το σενάριο φαίνεται απίθανο. Εκτός αυτού θα απαιτούσε και αναθεώρηση των συνθήκων για την διάκριση μεταξύ πολιτικού και στρατιωτικού. Τρίτο σενάριο, η ενδυνάμωση της Αθηνάς μέσω της διεύρυνσης, της επέκτασης των του κόστους που αναλαμβάνει. Ιδιαίτερα το κόστος μεταφοράς όπως τη μεταφορά των bell groups. Αλλά δεν υπάρχουν μόνο αυτά γιατί αυτά υποχρησιμοποιούνται. να υπάρξουν, να αναλάβει η Αθηνά πολύ μεγαλύτερο τμήμα του κοινού κόστους. Αυτό το σενάριο είναι πιθανό και αληθοφανές. Ναι, εάν οι διάφοροι παράγοντες λάβουν υπόψη τους όντως όλο το κόστος, αλλά η αναθεώρηση του κανονισμού της Αθηνάς που θα ολοκληρωνόταν θεωρητικά το Δεκέμβριο του 2014 φαίνεται δύσκολη. Υπέρ και κατά ένα μεγάλο υπέρ ότι θα χορηγούνταν περισσότεροι πόροι και θα γίνονταν οι επιχειρήσεις πολύ γρηγορότερα. Καθώς και μεγαλύτερη αλληλεγγύη αφού θα συμμετείχαν περισσότερα κράτη. Κατά, αν δεν περάσει όλο το κόστος στην Αθηνά, τότε παραμένει το πρόβλημα του κόστους που θα αναλαβουν μονομένα μεμονωμένα κράτη-μέλη. ως προς την ταχύτητα. Εδώ ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα κινητοποίησης, χρήσης των πόρων που διαθέτουν τα κράτη-μέλη, έξω και η ιδέα ενός startup fund που θα επέτρεπε την επιτάχυνση της λήψης των αποφάσεων και ιδίω της κινητοποίησης των πόρων. Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται από τις ηθίκες. Είναι εύκολο να εφαρμοστεί κατά ένα θέμα συνέπειας και συνοχής, γιατί αν δεν δυναμωθεί η Αθηνά θα υπάρξει μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ Αθηνάς και προϋπολογισμού. Και έπειτα η Αθηνά δεν δίνει καμία εγγύηση για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Παραμένει λοιπόν ένα τέταρτο σενάριο η προοδευτική συμπερίληψη όλου του κόστου στον προϋπολογισμό. της Ένωσης. Αυτό λέω προοδευτικά για να μην γίνει απότομα, αλλά μπορεί κανείς να φανταστεί ότι μερικές δαπάνες της Αθηνάς θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό, ενώ οι εθνικές εισφορές να παραμείνουν στην Αθηνά. Μία παράλληλη δηλαδή εξέλιξη προς την προοδευτική συμπερίληψη στον προϋπολογισμό. Τώρα, είναι πιθανό η αληθοφανές αυτό. Δεν ξέρω αν τα κράτη θα δεχτούν τέτοια μέτρα, αλλά μία πρώτη τέτοιου είδους εξέλιξη έγινε από το 1997 όταν αποφασίστηκε η αυτόματη χρηματοδότηση των πολιτικών επιχειρήσεων από τον προϋπολογισμό. Τα υπέρ θα ήταν μεγαλύτερη συνέπεια και συνοχή, περισσότερος δημοκρατικός έλεγχος και περισσότερη αλληλεγγύη. Αν και δεν υπάρχουν εδώ πλήρεις εγγυήσει, παρόλα αυτά είναι μια λύση που με βάση αυτά τα κριτήρια φαίνεται μάλλον σωστή. Τα κατά η ταχύτητα της ανάδρασης, αντίδρασης δεν είναι εγγυημένη γιατί όλα εξαρτώνται από την καλή θέληση των οργάνων και ούτε υπάρχει η εγγύηση ότι η συνολική πόρη θα είναι υψηλότερη για όλες αυτές τις επιχειρήσεις και αποστολές. Η κυριότερη δυσκολία είναι ότι και εδώ απαιτείται αναθεώρηση των συνθήκων λόγω της διαφοράς πολιτικής και στρατιωτικής δράσης. Τελειώνω τώρα λέγοντας ότι ε, πέρα από αυτά τα τέσσερα σενάρια Υπάρχουν δυνατότητες ενισχυμένης συνεργασίας με ορισμένων κρατών που προβλέπεται από τη συνθήκη η δυνατότητα μια ομάδας κρατών να εφαρμόσει μια επιχείρηση με βάση την έγκριση και των υπολείπων και η περίφημη μόνιμη και δομημένη συνεργασία. Ούτε αυτό βέβαια δεν λύνει το πρόβλημα της χρηματοδότησης στο σύνολό του, γιατί ακόμη και αν επιλεγόταν αυτή η λύση, θα έπρεπε να δούμε μετά πώς οι μηχανισμοί αυτοί συνεργασίας θα μπορούσαν να χρηματοδοτηθούν. Λέω απλώς ότι ερωτώ. Βλέπει κανείς, προβλέπει μεγαλύτερη αλληλεγγύη επειδή όλα τα κράτη θα έχουν δεχτεί ακόμα και αν ορισμένα μόνο αναλάβουν την επιχείρηση. Τέλος. Η εξέλιξη αυτών των δομών χρηματοδότησης εξαρτάται από τρεις, τρία είδη λογικής. Ο δισταγμός των χωρών μελών μήπως χάσουν τον έλεγχο των επιχειρήσεων. Η θέληση των θεσμικών οργάνων, υπερεθνικών θεσμικών οργάνων να προχωρήσουν όλα αυτά προς μεγαλύτερη ολοκλήρωση και τρίτον οι επιχειρησιακές ανάγκες της ΚΠΑΣΑ αν θέλουμε να παίξουμε ρόλο διεθνή. η ενίσχυση της ΚΠΑΣΑΘ σημαίνει πιο συλλογική χρηματοδότηση είτε με την ενδυνάμωση της Αθηνάς είτε μέσω μεγαλύτερης συμπερίληψης στον προϋπολογισμό. Αυτό μου φαίνεται απολύτως σαφές. Το θέμα όμως είναι αν όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα συμφωνήσουν η Κομισιόν, η Εξωτερική Υπηρεσία, η Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων, τα κράτη-μέλη αν πισθούν ότι οι ανάγκες της ΚΠΑΣΑ πρέπει να χρηματοδοτηθούν περισσότερο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε και εμείς ε, πολύ και ζητώ συγγνώμη για άλλη μια φορά που ε, δεν σας παρουσίασα σωστά στην αρχή. Έχουμε λοιπόν δύο εισηγητές. Ο κύριος Κούκαν θα λάβει το λόγο εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και επίσης ε, σας ευχαριστώ και για το ότι ε, καλέσατε τον καθηγητή κύριο Τέρπαν. Ακούσαμε μια πάρα πολύ σημαντική παρουσίαση ε, και μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν μια ομιλία που δεν μπήκε σε επιστημονικό αναλυτικό βάθος αλλά προσέγγισε το όλο θέμα κάτω από ρεαλιστικό πρίσμα που να μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε την ε, παρουσίασή του αυτή. Δεν είναι μια θεωρητική προσέγγιση, καθαρά πρακτική ήταν που αφορά άμεσα στο, στην έκθεση και στο ψήφισμα που προτιθέμεθα να υιοθετήσουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να αναφέρω ορισμένα θέματα που αφορούν στην έκθεση της ε, Επιτροπής μας. Πρώτον, ορισμένα γενικής φύσεως θέματα. Συζητάμε για αυτή την έκθεση όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει προκλήσεις ε, χωρίς προηγούμενο και πολλές απειλές ως προς την ασφαλειά της. Βεβαίως όλοι γνωρίζουμε την κατάσταση στην ε, γειτονιά μας ε, προς Ανατολάς, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές απειλές από τη Μέση Ανατολή και από την Ανατολική Αφρική. Για να αντιμετωπιστούν λοιπόν πολλές από αυτές τις προκλήσεις και να συνεχίσει να υπάρχει ασφάλεια, αυτή τη στιγμή έχουμε 17 στρατιωτικές και πολιτικές επιχειρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακάμπτει από την οικονομική κρίση που έχει πλήξει τις ε, δαπάνες και για την άμυνα. Τα περισσότερα κράτη-μέλη δεν ήταν πρόθυμα να διαθέσουν περισσότερους πόρους ε, ε, για την κοινή άμυνα και στον ε, προϋπολογισμό, ο προϋπολογισμός για την ε, άμυνα και την ασφάλεια υφίσταται μεγάλους περιορισμούς. Γι' αυτό λοιπόν καλούμεθα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μέσα σε αυτό αυτούς τους ε, περιορισμούς για την ΚΠΑ. Το βασικότερο είναι να εντοπίσουμε τα προβλήματα, να δούμε τι αποθέματα έχουμε και να προτείνουμε πιο αποτελεσματικούς αλλά και διαφανείς τρόπους για να χρηματοδοτήσουμε αυτή την πολιτική. Αυτά ήταν τα γενική φύσεως και τώρα θα περάσω στα πιο συγκεκριμένα. Όπως σας είπα, οι βασικές προκλήσεις για την έκθεση είναι να βρούμε πώς θα ταυτίσουμε τους περιορισμένους πόρους για την ΚΠΑ και τις νέες νέες φιλοδοξίες για την πολιτική μας. Πρέπει να αναλύσουμε τη ε, διαθεσιμότητα των οικονομικών πόρων και να υπογραμμίσουμε επίσης ε, την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών χρηματοδότησης και τη διαχείριση, τη σωστή διαχείριση των αποστολών στο πλαίσιο της ΚΠΑ. Νομίζω ότι αξίζει το κόπο να αναφέρουμε τους περιορισμούς που υπάρχουν κυρίως για τις πολιτικές αποστολές και ε, αυτό μας ανάγκασε να ε, μεταφέρουμε στο 2015 τους μη πληρωμένους λογαριασμούς σε τάξεις περίπου 30 δις ευρώ. Είναι εξίσου σημαντικό να ενισχύσουμε το δημοκρατικό έλεγχο και την ε, κοινοβουλευτική διάσταση της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Θα ήθελα στην έκθεση να γίνεται έκκληση στο να υπάρχει ξεχωριστή δημοσιονομική γραμμή στον προπολογισμό για κάθε επιχείρηση της ΚΠΑ, έτσι ώστε να υπάρχει και μεγαλύτερη διαφάνεια στη χρηματοδότηση των αποστολών. Όσον αφορά τη δομή της έκθεσης, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να εξετάσουμε τη δυνατότητα εξοικονόμησης δαπανών, να υπάρχουν ας πούμε κοινά κέντρα παροχής υπηρεσιών, αλλά εξοικονόμηση να υπάρχει και στις διαδικασίες δημόσιων διαγωνισμών. Επίσης θα έπρεπε να εξετάσουμε και το θέμα της ε, συνοχής και της ε, συμπληρωματικότητας των αποστολών της ΕΚΠΑ, ε, συμπληρωματικότητα και με άλλους οργανισμούς όπως είναι παραδείγματος χάρη το ΝΑΤΟ. Η χρηματοδότηση των στρατιωτικών αποστολών έχει σχέση με θέματα οικονομικής διαχείρισης των στρατιωτικών και των πολιτικών αποστολών. Και εδώ θέλω να εξετάσω το θέμα της αναθεώρησης του μηχανισμού Αθηνά. Αυτή βέβαια είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την έκθεση και με ενδιαφέρει πάρα πολύ η συζήτηση που θα ακολουθήσει για να έχω και εγώ κάποιες περισσότερες ε, προτάσεις και νομίζω ότι θα διαμορφωθούν περισσότερες απόψεις σχετικά με την έκθεση. Ε, και θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο καθηγητή. Όπως σας είπα, η έκθεσή του είναι πολύ σημαντική. Είναι πρακτικά, πρακτική, ρεαλιστική και συμφωνώ μαζί του όσον αφορά τον εντοπισμό των βασικότερων ε, προβλημάτων σχετικά με τη χρηματοδότηση της ΚΠΑ, όπως παρουσίασε ο ίδιος αυτά τα προβλήματα. Πράγματι δεν υπάρχει αποτελεσματικότητα, δεν υπάρχει δημοκρατία και διαφάνεια, αλλά δεν υπάρχει και αλληλεγγύη και αυτά αναχαιτίζουν την αποτελεσματική χρηματοδότηση και λειτουργία των επιχειρήσεων. Είναι σημαντικό να ακούσουμε διάφορες απόψεις ως προς και στα διαφορετικά ε, σενάρια για τη χρηματοδότηση. Το να διατηρηθεί το καθεστώς ως έχει, αυτό νομίζω μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Θεωρώ ότι σταδιακά θα πρέπει να περάσουμε σε αυτό ε, που αποκαλείται budgetization των ε, επιχειρήσεων ε, και με πολύ χαρά θα άκουγα τις απόψεις των συναδέλφων μου επ' αυτού. Μία τελευταία μου πρόταση. Ε, είναι σημαντικό να υπάρχει μεγαλύτερη πολιτική συνένεση για να πράξουν περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στην ΚΠΑ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Κούκαν. Αυτό το θέμα που εξετάζουμε είναι πάρα πολύ περίπλοκο και θα πρέπει να συζητηθεί και κάτω από το ε, πρίσμα της ε, χρηματοδότησης. Δίνω το λόγο στο δεύτερο εισηγητή, ο οποίος θα εκπροσωπεί στην Επιτροπή Προϋπολογισμών. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι μεγάλη τιμή και μεγάλη χαρά να μπορώ να συνεργάζομαι με την υποεπιτροπή σας, δίνοντάς σας την προσέγγιση της Επιτροπής Προϋπολογισμών που δεν είναι κατά ανάγκη αρνητική ή κακή. Απλά εμείς πιστεύουμε ότι η ΚΕΠΑ και η ΚΠΑ πρέπει να οργανωθούν πολύ καλύτερα σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο είναι αυτή τη στιγμή οργανωμένες. Έχω χωρίσει την παρουσίασή μου σε δύο μέρη. Το πρώτο είναι οι μη στρατιωτικέ επιχειρήσεις. Είδαμε ότι υπάρχουν ζητήματα με τη χρηματοδότησή του Ήδη όταν προδεκαετίας ξεκίνησε η πρώτη μη στρατιωτική επιχείρηση, το διαπιστώσαμε αυτό το πρόβλημα. Συνήθως τα προβλήματα έχουν να κάνουν με την διοικητική μέρημνα και τις υποδομές. Υπάρχει ένα επιχείρημα να αλλάξουν χρηματοδοτικοί κανόνες. Να υπάρχουν ειδικοί κανόνες δηλαδή για τις μη στρατιωτικέ επιχειρήσεις. Θεωρούν ορισμένοι ότι είναι δυνατόν να υπάρξει ταχύα ανάπτυξη εντός του υφιστάμενου πλαισίου, αλλά την απόφαση θα πρέπει να τη λάβουμε εμείς, καταρτίζοντας αυτή την έκθεση. Επίσης, τι θα γίνει με τη διαθεσιμότητα του εξοπλισμού. Αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εξοπλισμούς προηγούμενων αποστολών και νομίζω και από τον ΑΣΕ γίνεται κάτι ανάλογο. Σίγουρα ο ρόλος του μηχανισμού είναι σημαντικός και αυτό είναι το δεύτερο σκέλος μηχανισμό Αθηνά, όπως μας τον παρουσίασε ο εμπειρογνώμων μας, τον οποίο και ευχαριστώ, είναι σημαντικός και πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργεί πιο αποτελεσματικά στο μέλλον. Τα κράτη-μέλη βέβαια. Θα πρέπει να χρηματοδοτήσουν ε, την ανάπτυξη αυτών των δυνάμεων κυρίως από τον εθνικό τους προπολογισμό, εξού και η επιφυλακτικότητά τους. γιατί πετούνται διαφορετικές προσεγγίσεις ενίοτε. Αν κατάλαβα καλά, οι κοινέ δαπάνες, αντιεθνικών δηλαδή δαπανών, θεωρείται μια επιλογή που την ασπάζονται πολύ εδώ στο Κοινοβούλιο. Και ολοκληρώντας, να πω ότι και οι συναδελφοί της Επιτροπής ε, αλλά φαντάζομαι και υπό επιτροπή σας έτε, μπορούμε να συνεργαστούμε για να επηρεάσουμε την έκθεσή μας όσο το δυνατόν περισσότερο και να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Διότι πιστεύω ότι με τον τρόπο αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση τη δεσμεύση που ανέλαβε, το Συμβουλίο Θεσσαλονίκη, ε, τους ε, στόχους του Ελσίνκη, δήλωση Πέιτερσμπουργκ κτλ. κτλ. Άλλωστε έχουμε μια ειδική γεωγραφία που σχετίστηκε με την κοινή πολιτική άμυνας. Δεν την έχουμε ακόμη αναλάβει εξ ολοκλήρου αυτή τη δέσμευση. Αλλιώς και ο Πούτιν δεν θα είχε ποτέ καταλάβει την Κρυμαία. Thank ε, Σας ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ Έχουμε τώρα εκπροσώπους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Θα δώσω καταρχάς ε, το λόγο όμως ε, στον ε, κύριο Κένεθ Ντίν, που είναι ο επικεφαλής της μη στρατιωτικής δυνατότητας σχεδιασμού και διεξαγωγής επιχειρήσεων. PCC. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε δυνατότητα να συμμετάσχω σε αυτή τη συζήτηση η ΕΙΕΔ χαίρεται πολύ που μπορεί να συνεισφέρει από αυτό το πρώιμο στάδιο στην κατάρτιση της έκθεσης. Θα μιλήσω για τις μη επιχειρήσεις και κάποια κοινά μέτρα και μετά θα δώσω και το λόγο στο συνάδελφό μου από την Υπηρεσία για τα εργαλεία εξωτερικής πολιτικής. Το 2014 είχαμε υποβάλει ένα συνοπτικό έγγραφο για τις στρατιωτικές, μη στρατιωτικές επιχειρήσεις και τα συνοδευτικά μέτρα μετά τα πορίσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου 2013. Είναι ένα έγγραφο το οποίο είναι αυτή τη στιγμή στη φάση αναθεώρησης και εξέτασης στα κράτη-μέλη. Ε, μελετήσαμε 10 μυστιωτικές επιχειρήσεις, τρισυπήρους, 7 προτάσεις ε, σε σχέση με τέτοιες επιχειρήσεις. Δεν είχαν μεγάλο αντίκτυπο. Ο στόχος ήταν να έχουμε ε, περιθώρια οικονομικά για να μπορέσουμε ενδεχομένω να ξεκινήσουμε και νέε δράσει το 2015. Η ΕΕ συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διάφορα ζητήματα. Ε, στόχος μας είναι βέβαια να έχουμε ταχύτερη ανάπτυξη των μη στρατιωτικών επιχειρήσεων, αλλά να βελτιώσουμε και την χρηματοοικονομική διαχείριση αποστολών και επιχειρήσεων. Επίση νομική ικανότητα, πρόσβαση στον προπολογισμό, νέε διαδικασίε διαχείριση κρίσεων είναι δείγματα τη πρόοδου που έχουμε διεπιτύχει στον τομέα αυτό. Παραμένουν βέβαια ζητήματα στα οποία μπορούμε να έχουμε ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση, ανέφεραν ε, οι συγητές σχετικά η ιδέα, παραδείγματο χάρη, ε, της ε, υποστήριξης αυτών των ε, επιχειρήσεων και από την πλευρά της δίκης και από την πλευρά των δημοσίων προμηθειών. Θέλουμε να έχουμε επίσης ένα είδος πλατφόρμα στήριξης των επιχειρήσεων, πάλι με στόχο τη συγκέντρωση. Και σε ό,τι αφορά το καθεστώς των διεθνών εργολάβων. Θέλουμε να έχουμε συνεπείς ενεκτικούς κανόνες και σαφείς διαδικασίες για τις μη σταθιωτικές επιχειρήσεις ε, ΚΠΑ, σε ό,τι αφορά το προσωπικό. Έχουμε και διοργανική ε, συζήτηση για μεγαλύτερη ευελιξία σε ό,τι αφορά τους οικονομικούς κανόνες και τους ε, διαγωνισμούς προμήθειες. Τα είπα και προλαλήσαντες. Και σε ό,τι αφορά ακριβώ αυτό το σημείο των κανόνων για τις προμήθειες, η ΕΕΔ συνεχίζει να προωθεί βελτιώσει για να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία με βάση, όπως είπα, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2013. Περαιτέρω ευελιξία, περαιτέρω πρόοδος φυσικά και θα ήταν ευπρόσδεκτη. Ε, θέλουμε να ορίσουμε καλύτερα την έννοια της κρίσης σε ό,τι αφορά τις ε, μη στρατιωτικές επιχειρήσεις και να αντιμετωπίσουμε και συγκεκριμένες προτάσεις για να διευκολύνουμε ε, και την ε, πιο ε, πρόημη και αποτελεσματική δρομολόγηση των διαδικασιών δημοσίων προμηθειών. Έχουν αναφερθεί κάποια καλά παραδείγματα πρόοδου, που νομίζω όμως ότι μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Πρόσβαση, καταλληλότητα, διαθεσιμότητα άρα συνεχίζουμε να δουλεύουμε. Έρχομαι στρατιωτικές επιχειρήσεις και τα συνοδευτικά μέτρα. Ήδη ο καθηγητής ε, Τέρπαν και οι συγητές έκαναν κάποια σχόλια. Δεν χρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό όπως προβλέπει η συνθήκη, χρηματοδοτούνται από τα μεμονωμένα κράτη-μέλη. Το λέει ο κανόνας, το άρθρο, το ε, αντίστοιχο τη συνθήκη, αυτά δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Τα είδαμε και στην παρουσίαση. Αυτή τη στιγμή έχουμε έξι στρατιωτικές επιχειρήσεις, μία στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, 19 Γενάρη ξεκίνησε, 85 εκατομμύρια ευρώ είναι το κοινό στρατιωτικέ επιχειρήσει. μια στην κεντροαφρικανικη δημοκρατια 19 γεναρη ξεκινησε 85 εκατομμυρια ευρω το κοινο κοστος των εξι στρατιωτικων επιχειρησεων και εκεί υπήρχε μια παράγραφος ε, ειδικά για τον αναθεωριστό μηχανισμό Αθηνά. Γιατί υπάρχουν κάποια ζητήματα που ενδιαφέρουν τα κράτη-μέλη και έχουν να κάνουν με την εφαρμογή και την εντολή. Για να δούμε πώς μπορεί να είναι πιο ευέλικτες κάποιες διατάξεις και διαδικασίες. Σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση του μηχανισμού. Δεν έχουμε ακόμη επίσημη έγκριση γιατί δεν υπάρχει εντολή από τα κράτη-μέλη για να ολοκληρώσουμε, να δυστυχοποιήσουμε αυτό το ζήτημα, σε ό,τι αφορά το κόστος ανάπτυξη των μάχημων ομάδων, των battle groups. Τα είπε ο καθηγητής. Ε, συντομία για το άρθρο 44 της συνθήκης, για τα συνοδευτικά μέτρα, να πω κάτι, είναι ένα άνθρωπο που δίνει τη δυνατότητα να ε, ανατεθεί ένα καθήκον ΚΠΑ σε μια ομάδα κράτων μελών μάλλον σε ό,τι αφορά τι αποστολέ ΠΑ. τώρα το Συμβούλιο εξετάζει το ενδεχόμενο αυτό να γίνεται και για αποστολέ και επιχειρήσει ΚΠΑ. Δεν θέλουμε όμως ε, να υποκαταστήσει το άρθρο αυτό την ε, πρότυπη έγκριση, αδειοδότηση ε, για την ανάπτυξη στρατιωτικών και επιχειρήσεων. Σε αυτή τη φάση τουλάχιστον. Θα μπορούσε όμως να χρησιμοποιηθεί κυρίως για τις στρατιωτικές και όχι για τις μη στρατιωτικές επιχειρήσεις είναι θέμα ερμηνεία των κρατών μελών και του Συμβουλίου. Μία επιλογή θα ήταν ε, οι ανθρωπιστικές επιχειρήσεις. Τέλος, ένα σημαντικό στοιχείο. Συνέργειες μεταξύ στρατιωτικών και μη στρατιωτικών μέσων. Δηλαδή, να αναπτύξουμε τους σωστούς ανθρώπους στο σωστό χρόνο, στο σωστό τόπο για να αντιμετωπίσουν τις σωστές ανάγκες. Να έχουμε λοιπόν συνεργασίες, ε, συγκέντρωση των δυνάμεών μας για να αντιμετωπίζουμε τις εκάστοτε ανάγκες ε, όπου και όποτε προκύπτουν. Θέλουμε να είμαστε πιο αποδοτικοί, πιο αποτελεσματικοί ε, στις στρατιωτικές μη στρατιωτικές επιχειρήσεις, ιδίως όταν έχουμε το ίδιο θέατρο επιχειρήσεων, Μάλι, Σομαλία, ίσως στο μέλλον και την Αφρικανική Δημοκρατία κόστος υπάρχει βέβαια. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάποια εξοικονόμηση αν είχαμε αυτές τις κοινέ επιχειρήσεις στρατιωτικών και στρατιωτικών. Θέλουμε να είναι ασφαλής ε, και η μη στρατιωτική αξιωματούχοι όταν αυτοί μεταβαίνουν σε κάποιες περιοχές για να εκτελέσουν ε, τα καθηκοντά τους. Αυτά λοιπόν τα πράγματα, όπως είπα, μας περιορίζει η συνθήκη, αυτά προβλέπει, αυτά μπορούμε να κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο. Uh, of the Commission. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γκάμιλα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πρόεδρε και συμπρόεδρε. Όπως αναφέρθηκε, εγώ ασχολούμαι ε, με την εξωτερική πολιτική, την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και συνεργάζομαι με τον συνάδελφό μου υπό την κυρία Μογκερίνη. Ε, και εμείς θέλουμε να καλωσορίσουμε την ε, πρωτοβουλή σας για την κοινή αυτή συζήτηση που λαμβάνει η χώρα σήμερα. Με χαρά περιμένω το σχέδιο της έκθεσης ε, και αυτή τη στιγμή βέβαια είναι δύσκολο να μπούμε σε λεπτομέρειες αλλά εν ευθέτω χρόνο θα δώσουμε και εμείς τη δική μας άποψη για τη δουλειά σας. Εγώ θα περιοριστώ σε κάποια γενικής φύσεως ε, θέματα. Θα κάνω δύο γενικής φύσεως παρατηρήσεις. Μία αφορά στον ε, προϋπολογισμό, ε, στην ΚΠΑ και στην ΚΕΠΑ μάλλον και πώς ακριβώς εφαρμόζεται ο προϋπολογισμός. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να επενθυμίσουμε τις παραμέτρους ε, μέσα ε, στις οποίες λειτουργεί ο προϋπολογισμός της ε, ΚΕΠΑ. Ορισμένα αναφέρθηκαν από τον εισηγητή ή τους εισηγητές και τον καθηγητή. Ο προϋπολογισμός της ΚΕΠΑ καλύπτει μόνο μη στρατιωτικές αποστολές της ΚΕΠΑ. Οι στρατιωτικές αποστολές με αμυντικές προεκτάσεις προφανώς δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τον προπολογισμό με βάση τις συνθήκες. Και για να γίνει κάτι τέτοιο όμως θα έπρεπε να αλλάξουν οι συνθήκες όπως είπε και ο κύριος καθηγητής. Βέβαια στην Επιτροπή και όχι μόνο στο FBI ε, προσπαθούμε να αναζητήσουμε την ε, συμπληρωματικότητα, τα συνοδευτικά μέτρα και όλα τα άλλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η δική μας η προσέγγιση αφορά στο να διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια ολιστική προσέγγιση. Όσον αφορά τώρα τις ε, χρηματοδοτικές ε, παραμέτρους, ε, νομίζω ότι είναι σαφής το επίπεδο του προεπλισμού για την ΚΕΠΑ έχει συμφωνηθεί στο πλαίσιο του πολιτούς δημοσιονομικού πλαισίου μέχρι το 2020. Έχει συμφωνηθεί περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ είναι το ποσό ε, προσαρμοζόμενο στον πληθωρισμό αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο δουλεύουμε και αυτό είναι ο προπολογισμό που υπάρχει στη διάθεσή μα. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι το Συμβούλιο και τα κράτη-μέλη αποφασίζουν επί των δράσεων που θα αναπτυχθούν ε, και επί του περιεχομένου των επιχειρήσεων. Αυτό είναι σημαντικό να το υπενθυμίσουμε. Στο πλαίσιο τη εξωτερική ε, πολιτική ε, προσπαθούμε να έχουμε έναν αποτελεσματικό προπολογισμό ε, τα μέλη της Επιτροπής ε, γνωρίζουν ότι αφήνουμε και ένα περιθώριο για πρόβλεπτα γεγονότα. Το 2015 υπάρχουν πολλές ε, δράσεις που συνεχίζονται. Οι γραμμές του προπολογισμού θα εξαντληθούν, αλλά νομίζω ότι και φέτος θα πρέπει να αφήσουμε ένα ικανοποιητικό περιθώριο για νέες δράσεις ε, που θα κληθούμε να χρηματοδοτήσουμε συζητήσουμε αν τελικά αναπτυχθούν δύο νέες επιχειρήσεις, αν κριθεί κάτι τέτοιο απαραίτητο. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, αν κριθεί πολιτικά απαραίτητο, πάντα υπάρχει δυνατότητα να ζητήσει κανείς περισσότερα κονδύλια. Και δεν νομίζω ότι χρειάζεται αυτό να το επαναλάβω ενώπιον της Επιτροπής Προϋπολογισμών, ότι υπάρχουν διάφορες τεχνικές για να το κάνει κανείς αυτό. Σε τελική ανάλυση, βεβαίως, η απόφαση είναι πολιτική, είναι η αρχή του προεπλογισμού του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου που αποφασίζουν επ' αυτών των θεμάτων. Όσον αφορά λοιπόν στην ε, εφαρμογή όλων αυτών και από αυτά που ελέγχθησαν, η Επιτροπή συμφωνεί απόλυτα με αυτά που ελέγχθησαν για την αποτελεσματική εφαρμογή της ε, ΚΕΠΑ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κοινή Εξωτερική Πολιτική και άλλες ε, υπηρεσίες συνεργάζονται στενά για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τις αποφάσεις του Συμβουλίου του 2013. Και εγώ ε, θα συνεχίσω να συνεργάζομαι με τους συναδέλφους μου. Ε, αναφέρθηκε και η ιδέα ενός ε, κέντρου. Υπάρχει αυτή η ιδέα εδώ και καιρό. Η Κομισιόν έχει διεξάγει μια μελέτη σκοπιμότητας για διάφορες συνέργειες, ε, μελέτη κόστους ωφέλους. Εμείς ε, στηρίζουμε πρωτοβουλίες προς αυτήν την ε, κατεύθυνση. Θεωρούμε ότι είναι ελπιδοφόρες για το μέλλον, γιατί το περιβάλλον μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας είναι αρκετά περίπλοκο, αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι θα βρεθούν κάποιες λύσεις. Και αυτή τη στιγμή εργαζόμεθα επί των λεπτομεριών. Όπως αναφέρθηκε, συνεχίζονται εργασίες για να υπάρχει μια κοινή πλατφόρμα και στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή θα μας επιτρέψει να εξορθολογήσουμε καλύτερα τα υπάρχοντα κονδύλια για να στηρίζουμε καλύτερα και τις επιχειρήσεις που αναπτύσσονται. Να τις απαλλάξουμε από το βάρος που τις επιβαρύνει κυρίως σε διοικητικό επίπεδο, κυρίως κατά τη φάση της ε, σύστασης. Αναφέρθηκε και το θέμα του Warhouse Το που έχει σημασία είναι ότι επ' αυτού ε, θα πρέπει να λειτουργήσουμε πριν το Συμβούλιο λάβει μία απόφαση. Τελειώνοντας ε, λοιπόν, ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα στηρίξει αυτήν την ε, πρωτοβουλία από κοινού με τους συναδέλφους από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Προφανώς και είμαστε πρόθυμοι να στηρίξουμε τους ηγητές, να τους ενημερώσουμε λεπτομερώς για το τι ακριβώς κάνουμε και είμαστε βεβαίως ε, και στη διάθεση όλων των μελών και των δύο επιτροπών αν χρειάζονται τις ε, πληροφορίες μας και την υποστήριξή μας για να προχωρήσουν τη δουλειά Ξεκινάει λοιπόν η συζήτηση. Καταρχήν ο κύριος Γκάλα από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ τον ε, καθηγητή εισηγητή, τον δικό μας τον εισηγητή και επίσης και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Βεβαίως ε, τα ε, σημεία κίνησης των σκέψεών μας είναι οι υπάρχουσες συνθήκες. Πάνω σε αυτές βασιζόμαστε. Ακόμα και αν επιθυμώ να υπάρξει μια νέα συνθήκη, να εξευρετούν ε, νέοι μηχανισμοί. Γιατί μεταξύ άλλων αναφέρθηκε το ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει αυτός ο τεχνητός διαχωρισμός ανάμεσα στις μη στρατιωτικές και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Δεν διαχωρίζονται πλήρως, ε, αλλά επειδή υπάρχουν κάποια τέτοια στοιχεία, μη στρατιωτικά και στρατιωτικά, τα πράγματα δυσκολεύονται με τη χρηματοδότηση. Βεβαίως ε, είναι γνωστό και το πρόβλημα που υπάρχει στις εφαρμόσιμες ε, πρακτικές, ε, στη χρηματοδότηση, στον ε, τομέα των μη στρατιωτικών επιχειρήσεων. Οι συνάδελφοι αναφέρθηκαν λεπτομερώς που ακριβώς βρίσκονται τα πρακτικής φύσεως προβλήματα. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα το οποίο για μένα είναι πρωταρχικής ε, σημασίας. Είναι το εξής, αυτό το μηχανισμό Αθηνά, πώς μπορούμε να τον μεταρρυθμίσουμε προς όφελος των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Να πω το εξής, καταρχήν, ό,τι γίνεται σε αυτόν τον τομέα ε, έχει αποφασιστεί ομόφωνα. Αυτό είναι ευχάριστο. Άρα δηλαδή μπορεί κανείς να θεωρεί ότι όλα τα κράτη-μέλη δεσμεύονται από κοινού για μια κοινή υπόθεση. Και κατά την άποψή μου από εκεί απορρέει και το δεύτερο βήμα ότι δηλαδή αυτή η κοινή ανάληψη ευθυνών χρηματοδοτείται και από κοινού. Η πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε είναι αυτή που περιγράφηκε. Δηλαδή, πολύ λίγοι είναι εκείνοι οι οποίοι δυστυχώς πολλές φορές επιθυμούν να συνεργαστούν και όσο βέβαια πιο συχνά συνεργάζονται, τόσο πιο πολύ κατ' ουσίαν καλύπτουν μόνοι τους το κόστος. Το δικό μου λοιπόν το επιχείρημα απέναντι σε εκείνους οι οποίοι διαφωνούν, που δεν θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό το, στην κοινή ανάληψη ε, των ε, δαπανών, εγώ τους λέω ότι όποιος δεν το θέλει, αυτός ε, καλείται τις περισσότερες φορές να αναλάβει την ευθύνη και αυτό βεβαίως αφορά περισσότερο τα μεγάλα κράτη-μέλη. Γιατί υπάρχει μια κατάσταση όπου τα μικρότερα κράτη-μέλη που θα μπορούσαν να διαθέσουν ε, την υποδομή και τους ε, στρατιώτες δεν θέλουν να το κάνουν αυτό γιατί δεν μπορούν να αναλάβουν μόνα τους ε, το κόστος τα 100%. Μπορούν να συνεισφέρουν, να συνδράμουν στον κοινωνικό προπολογισμό αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν εξ ολοκλήρου το κόστος και γι' αυτό δεν συμμετέχουν. Αλλά λέει τι γίνεται τελικά. Τελικά παραμένουν εκείνοι που μπορούν να λάβουν το κόστος. Η συζήτηση λοιπόν στο Συμβούλιο θα πρέπει να είναι προς αυτή την κατεύθυνση από κοινού πράγματα που έχουν αποφασιστεί, μα από κοινού να χρηματοδοτούνται αυτά στο πλαίσιο της διαδικασίας που ισχύει, γιατί στη τελική ανάλυση συμβαίνει το εξής. Έτσι κι αλλιώς καταβάλει κανείς τη συνδρομή του που ε, προβλέπεται να καταβάλει αλλά δεν αναλαμβάνει ευθύνη. Αυτή τη λογική προσπαθώ εγώ να εξηγήσω στη Γερμανία και ελπίζω αυτό το θέμα να συζητηθεί και σε άλλες χώρες έτσι ώστε τελικά να μπορέσουμε να έχουμε πιο αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεών μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Mr. Munger, uh, but... Ο κύριος Μάγκα από την Επιτροπή Προεπλογισμών των Εκπροσωπών της Σοσιαλδημοκράτες. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν λοιπόν ε, τα κράτη-μέλη επιθυμούν να συνεργαστούν, εμείς πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό ε, θα μειωθεί η συνδρομή τους, ε, θα είναι μικρότερη από ό,τι είναι τώρα. Εγώ δεν είμαι εμπειρογνώμονας ε, για θέματα άμυνας, αλλά πιστεύω ότι με κοινή πολιτική μπορούμε να εξοικονομήσουμε πάνω από 26 δις, τα οποία μπορούμε να διαθέσουμε για άλλες επιχειρήσεις ή για άλλες πολιτικές. Ε, στον τομέα αυτό υπάρχουν ε, δυνατότητες βελτίωσης, να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, μεγαλύτερη διαφάνεια στις κρατικές προμήθειες, να υπάρχει ε, κοινός ε, χάρτη πορεία, ε, κάποια ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Υπάρχουν πολλά θέματα που καλούμεθα να εξετάσουμε και νομίζω με τον τρόπο αυτό θα μπορούμε να διαθέσουμε περισσότερα κονδύλια για την ασφάλεια μας. Ο κύριος Γερουσέμκο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για το ότι, κυρία Πρόεδρε, βάλατε αυτό το σημαντικό θέμα στην ημερήσια διάταξη. Και εγώ συνεχίζω εκεί που σταμάτησε ο προλαλής σας. Κατά τη δική μου λοιπόν άποψη αντιμετωπίζουμε ένα μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τη μεθοδολογία. Και παρακαλώ πολύ να λάβετε υπόψη στο εξή. Το θέμα με το οποίο ασχολούμεθα σήμερα είναι η χρηματοδότηση της ε, ΚΕΠΑ, της κοινή Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας. Και θέλω να σας επισημάνω το εξής. Εδώ στην Επιτροπή μας το γεγονός ότι ασχολούμεθα με την ΚΕΠΑ σημαίνει ότι ασχολούμεθα με την άμυνα. Και όταν πρόκειται για την άμυνα, κατ' ουσίαν πρόκειται για κοινέ επιχειρήσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά κατά πόσον η προσέγγιση μας ως προς αυτά τα θέματα δεν θα πρέπει να διευρυνθεί. Σήμερα μιλάμε για την ασφάλεια και συμφωνώ απόλυτα με τους ε, συναδέλφους ότι στην Ευρώπη αντιμετωπίζουμε τρομοκρατικές απειλές, προβλήματα με τη μετανάστευση, προβλήματα επίσης ε, με το ενδεχόμενο επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Άρα όλα αυτά τα προβλήματα πρέπει να τα εξετάσουμε εφόσον επιθυμούμε να ασχοληθούμε με την ανάλυση των δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της ασφάλειας. Είναι λοιπόν σημαντικό να περάσουμε και πέρα από τα αυστηρά όρια της άμυνας. Σημαντική είναι η άμυνα, αλλά η άμυνα είναι ένα κομμάτι, ένα σκέλος που έχει επιπτώσει στην ασφάλεια. Αυτά ήταν το πρώτο. Το δεύτερο που θέλω να πω, όλες οι εισηγήσεις μέχρι τώρα ήταν πολύ ενδιαφέρουσες, όμως ε, θέλω να παρατηρήσω το εξής. Το θέμα είναι ότι υπάρχει δυστυχώς μία πολύ χαλαρή προσέγγιση ε, Υπάρχει μια χαλαρή προσέγγιση ότι έχουμε μια σειρά κρατών ε, που λαμβάνουν αυτό το θέμα πάρα πολύ σοβαρά και που ε, χρησιμοποιούν δικά τους ε, κονδύλια για τις επιχειρήσεις, αλλά έχουμε και μια άλλη σειρά κρατών που δεν ε, συμβάλλουν καθόλου προς αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας στο θέμα αυτό. Πράγματι νομίζω ότι μπορούμε να διαθέσουμε τις πληροφορίες αυτές και στην, στα μέλη της υποεπιτροπής μας και στην Επιτροπή Προϋπολογισμών πριν την πρώτη εξέταση της έκθεσης. Θα δώσω τώρα το λόγο στον Αντιπρόεδρο της Υποεπιτροπής τον κύριο Χέλλερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή Ταπά για τη μελέτη που μας παρουσίασε γιατί με ιδιαίτερα ευκρινή τρόπο ε, παρουσιάζει ε, τα ελλείμματα και τα προβλήματα. Σπάνιο αυτό. Ε, μας παρουσιάζουν όλοι πολλά προβλήματα, αλλά εδώ κατέστη σαφές και το τι ακριβώς πρέπει να γίνει και ποια είναι τα υπέρ και τα κατά των επιλογών. Πολύ σύντομα θα ήθελα να ε, στις, ε, στο μη στρατιωτικό τομέα, να ευχαριστήσω θερμά τους εισηγητές, κυρίως ε, τους συναδέλφους της Επιτροπής Προπολογισμών και πάνω απ' όλα τον πρόεδρό τους. Νομίζω λοιπόν ότι η έκθεση έχει δύο πτυχές αναγκαστικά, γιατί βασιζόμαστε στις συνθήκες, αλλά δηλαδή υπάρχει καταρχήν ένα στοιχείο έκκλησης. Υπάρχει ο μηχανισμός Αθηνά, υπάρχει η προοπτική ε, των μη στρατιωτικών ε, επιχειρήσεων και εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να επιδεικνύουμε μία συνέπεια. Και υπάρχει ένα δεύτερο σκέλος που αφορά και βασίζεται στα άρθρα της ε, συνθήκης και εκχωρεί αυτό το σκέλος κάποιες αρμοδιότητες και κάποια επιρροή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό το σκέλος είναι ε, το μη στρατιωτικό. Και στα δύο σκέλη πρέπει να είμαστε σαφείς. Στο μη στρατιωτικό σκέλος πρέπει να πούμε με σαφήνεια ότι θέλουμε να υπάρχουν επιχειρήσεις που να μπορούμε να τις ε, διαχειριστούμε, που είναι ένα ουσιαστικό πολιτικό εργαλείο που ε, εκφράζουν και ταυτίζονται με ε, διεθνή πρότυπα, να υπάρχουν ε, οι διαγωνισμοί και εκδοτικές προσμήθειε και όλα αυτά να μπορούν να καλυφθούν από τον προϋπολογισμό. Επίσης να πούμε ότι οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν και την δική τους την αυτονομία στη χρηματοδότηση. Δεν είναι δυνατόν ο επικεφαλής μιας επιχείρησης να μην έχει το δικό του τον προϋπολογισμό. Βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη τους δημοσιονομικούς κανονισμούς και τον έλεγχο του προϋπολογισμού, αλλά όσο έχει τώρα το σύστημα δεν είναι μόνο αναποτελεσματικό, αλλά είναι και επικίνδυνο, πολύ επικίνδυνο. Υπάρχει ε, κάποιος κίνδυνος ελοχεύει κίνδυνο για την εξωτερική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι μόνο θέμα χρόνου ότι κάποια στιγμή κάποιο ε, στο πλαίσιο των ε, μη στρατιωτικών επιχειρήσεων θα υψώσει το ε, δάκτυλο σε ένα από τα κράτη-μέλη και θα πει ότι εμείς δεν θέλουμε να συμμετάσχουμε σε αυτήν την επιχείρηση γιατί είναι καθαρά ε, πολιτική, είναι στρατιωτική, μη στρατιωτική, δεν είναι αποτελεσματική. Άρα δηλαδή εδώ μιλάμε όχι μόνο για τα τεχνικά στοιχεία των ε, θεμάτων αλλά συζητάμε και για το κατά πόσο με το ισχύον καθεστώ η αξιοπιστία αυτών που κάνουμε στο πλαίσιο της ΚΕΠΑ η αξιοπιστία ισχύει ή όχι. Αυτό λοιπόν Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε το συντομότερο δυνατόν, γιατί αλλιώς σε αυτούς τους χαλεπούς καιρούς ο κύριος Πούτιν αλλά και άλλοι ε, θα καταλήξουν στην απάντηση ότι είμαστε τίγρης χωρίς δόντια, που δεν έχουμε καν τη δυνατότητα ακόμα και επιχειρήσεις που έχουν αποφασιστεί από τα κράτη-μέλη να εκτελούνται με αποτελεσματικότητα. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ, ναι μεν συζητήσαμε για πολλά από αυτά τα θέματα, αλλά θα πρέπει να συμφωνήσουμε πάνω σε σαφή σενάρια. Να περιγράψουμε με σαφήνεια το πώς θα λειτουργούν στο μέλος οι μη στρατιωτικές επιχειρήσεις. Και να εξηγήσουμε ποια είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον ε, θέμα του, ε, στο θέμα μηχανισμός Αθηνά. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ήμουν τόσο βέβαια για τους εκπροσώπους των συντηρητικών ποιος ήθελε να λάβει το λόγο. Άλλοι από τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον καθηγητή για την παρουσίασή του διότι μας περιέγραψε την πραγματική κατάσταση που ισχύει και γι' αυτό θα ήθελα να του θέσω δύο ερωτήματα για την κοινή πολιτική ασφαλείας κλπ. Άμυνας. Καταρχήν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Νοεμβρίου λένε ότι το Συμβούλιο δέχεται τα συμπεράσματα της τελευταίας διάσκεψης του ΝΑΤΟ όπου γίνεται συγκεκριμένα λόγος για την ανατροπή της τάσης μείωσης των προϋπολογισμών άμυνας. Γίνεται επίσης λόγος για πιο ισορροπημένη κατανομή και ζητιέται η ατήρηση ισχυρής αμυντικής βιομηχανίας και στην Ευρώπη και στα ΗΠΑ. Μερικοί ζήτησαν να μην μειωθούν οι στρατιωτικοί προπολογισμοί κάτω από, το 2, κάτω από 2%. Και η έρευνα για τα θέματα της άμυνας ε, να μην είναι χαμηλότερη από 20%. Πώς μπορούν όλα αυτά να μεταφραστούν στην, με όρους της ΚΠΑΣΑ. Τίθεται και το ερώτημα αν χρειάζεται αναθεώρηση των συνθήκων. Δεύτερον, το Συμβούλιο τονίζει ότι πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματική εκπάσα και άρα να, έχουν, παίζουν μεγαλύτερο ρόλο στις εισφορές τα κράτη-μέλη πράγμα που, πρέπει να θα μπορούσε να δημιουργήσει και περισσότερες θέσεις ασφαλείας λόγω της θέσης για την έρευνα και τη βιομηχανία. ο συντονισμός που γίνεται στην Ένωση υποστηρίζει άραγε αυτά τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Ο συντονιστής κύριος Φλόζινγκ της Γκουε. Ή κυρία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το θέμα είναι ιδιαίτερα περίπλοκο και ευχαριστώ θερμά ε, για την παρουσίαση του κυρίου καθηγητή ο οποίος ε, παρουσίασε με εύγλωτο τρόπο τα υπέρ και τα κατά. Εγώ ε, θα συνοψίσω αυτά που έχουν λεχθεί κατά το παρελθόν λέγοντας τα εξής, ότι πρέπει να διατίθενται περισσότερα κονδύλια για τον τομέα της ασφάλειας ε, ή για το στρατιωτικό τομέα, ότι δηλαδή έχει παρουσιαστεί η ανάγκη να διατίθενται περισσότερα κονδύλια σε αυτό τον τομέα. Ο άλλος τομέας περιγράφεται με εκφράσεις όπως ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και ούτω καθεξής. Βεβαίως ε, το υπόβαθρο πάνω στο οποίο στηρίζονται όλα αυτά παρουσιάστηκε από τους ομιλητές. Το υπόβαθρο είναι οι ε, συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω ο κύριος Γκάλα κατέστησε απόλυτα σαφές ότι κατ' ουσίαν ε, θα πρέπει να τροποποιηθούν αυτές οι συνθήκες. Και εδώ θέλω να σας πω ότι η δική μου η πολιτική ομάδα τάσεται κατά της τροποποίησης των συνθήκων για αυτό το θέμα. Ο κύριος Γκάλε έχει επίσης και το πρόβλημα ε, του διαχωρισμού ε, στρατιωτικού και μη στρατιωτικού. Αν κατάλαβα καλά, είπε ότι υπάρχει μια, ένας τεχνητός διαχωρισμός ανάμεσα στα δύο. Εμείς όμως είμαστε υπέρ του να υπάρχει μεγαλύτερος διαχωρισμός ανάμεσα στο, στις στρατιωτικές και μη στρατιωτικές επιχειρήσεις. Γιατί αλλιώς ε, πραγματικά θα ήταν μια τεράστια ανατροπή. Και εγώ έρχομαι στο στοιχείο του δημοκρατικού ελέγχου. Πιστεύω ότι με το να είναι ασαφή τα όρια είναι πολύ πιο δύσκολο να υπάρχει δημοκρατικός έλεγχος. Τα κράτη-μέλη στην τελική ανάλυση κανείς δεν θα ξέρει κατά πόσον πρόκειται για μια στρατιωτική ή μη στρατιωτική επιχείρηση. Η δυνατότητα των κρατών μελών να ε, συμμετέχουν, τέτοιο αυτό το θέμα, συζητήθηκε. Νομίζω λοιπόν ότι ε, το πρόβλημα ή το θέμα παρουσιάζεται ως πρόβλημα, αλλά εγώ ξέρετε το βρίσκω θετικό το ότι τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα στο πλαίσιο της ε, ε κυριαρχίας τους ε, σε θέματα προεπλισμού να αποφασίζουν μόνα τους που θα δαπανίσουν τα χρήματα και που όχι. Εγώ το βρίσκω σημαντικό να μπορούν να αποφασίσουν μόνα τους τα κράτη-μέλη στο μέλλον σε ποιες ε, στρατιωτικές επιχειρήσεις επιθυμούν να συμμετέχουν και σε ποιες όχι. Αυτή η δυνατότητά τους να διαφυλαχθεί, να παραμείνει και στο μέλλον. Ε, Λέχθησαν πάρα πολλά σχετικά με το ότι ο προϋπολογισμός ε, θα πρέπει να εξετάζεται κάτω από το πρίσμα των ε, ευρωπαϊκών, των ε, ενωσιακών δράσεων. Κάποιος μίλησε για το να διατίθεται κονδύλια για την έρευνα από τον προβλησμό. Επ' αυτό έχουμε συζητήσει τις συζητήσει εδώ στην Επιτροπή μας και διαφωνούμε, δίστανται οι απόψεις. Εγώ θα ήθελα να απευθυντώ στους εμπειρογνώμονες. Εκείνοι να μας πούνε ποια είναι τα ε, προκαταρκτικά μέτρα τα οποία ε, θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από τον προεπλογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, ποιες είναι τελικά αυτές οι στρατιωτικές δαπάνες. Το άρθρο 41 λέει ότι βασικά θέματα αποφασίζονται μόνο από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Εγώ αυτό το θεωρώ ότι είναι πρόβλημα. Είναι και ένα πρόβλημα που έχει να κάνει με τη συναπόφαση. Άλλο θέμα. Σχετικά με την έρευνα για τους εξοπλισμούς. Γίνεται μια συζήτηση από το Ταμείο να ε, χρηματοδοτούνται, να χρηματοδοτεί η έρευνα για τους εξοπλισμούς. Και συζητιέται επίσης κατά πόσον αυτό απαγορεύεται από το άρθρο 41.2. Αυτή την, αυτό το άρθρο το 41.2 εγώ το ερμηνεύω έτσι, ότι απαγορεύεται. Στο πλαίσιο των κείμενων συνθήκων καταβάλλονται διάφορες προσπάθειες να επικρατήσουν άλλες ερμηνείες. Αυτό όμως σημαίνει τροποποίηση των συνθήκων και γι' αυτό εγώ λέω να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια. Thank you. Uh, Madam uh, coordinator of Greens, SEDE. Συντονίστρια των Πρασίνων τη ΣΕΔΕ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεν έχω να προσθέσω πολλά σε όσα είπαν οι συνάδελφοί μου. Είπε κάποια πράγματα ο κύριος Γκάλε νωρίτερα όμως. Έκανε μια διάκριση μεταξύ μη στρατιωτικών και στρατιωτικών αποστολών και πρέπει νομίζω να μπει μια σαφή ή να διατηρηθεί αν θέλετε η σαφής διαχωριστική τραμμή μεταξύ των δύο. Γιατί αν τα αναμίξουμε θα δημιουργήσουμε προβλήματα περισσότερο τουλάχιστον από ό,τι ωφέλει. Σε πολλές περιπτώσεις το θέμα είναι οικονομικό. Δεν υπάρχουν χρήματα για παρέμβαση σε διάφορες χώρες. Έξω και δεν συμμετέχουν οι χώρες. Η Σουηδία, η χώρα μου, συχνά συμμετέχει σε αποστολές στατιοτικές και μη. Αλλά υπάρχει μια σαφής διάκριση. Ορίζουμε δηλαδή που μπορούμε να προσφέρουμε κάτι ώστε να είναι χρήσιμη η δική μας συμβολή στην κοινή επιχείρηση. Δεν είναι ίσως τόσο το οικονομικό, αλλά τι όφελος μπορεί να αποκομίσει μια κοινή επιχείρηση από τη συμμετοχή της Σουηδίας. Υπάρχουν χώρες που λαμβάνουν την απόφαση κάποιες φορές να μην συμμετάσχουν. Το θέμα είναι να κρίνουμε βάσει το όφελος. Thank you very much, uh, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, ο βασικός ε, στόχος είναι η επιτεύξη στρατηγικής αυτονομίας, δεδηλωμένα επίπεδα φιλοδοξίας της ΚΕΠΑ δεν ευθυγραμμίζονται με τις δυνατότητες και τον αμυντικό προπολογισμό των χωρών. Βλέπουμε ότι υπάρχουν διαφορετικές ελλείψεις και αυτό το βλέπουμε για αρκετά χρόνια τώρα. Και βέβαια λόγος είναι η οικονομική κρίση. Οι διαδικασίες λοιπόν αποφάσεων είναι μακροχρόνιες. Έχουμε αδράνεια στον τομέα της διοικητικής μέρημνης. Πρέπει όμως να χρηματοδοτηθούν σωστά οι αποστολές και οι επιχειρήσεις της Ένωσης. Αυτό είναι σημαντικό αν θέλουμε να έχει πραγματικό μέλλον η ΕΚΠΑ. Θα ήθελα λοιπόν να, να χαιρετήσω τη δημιουργία αυτού του κοινού κέντρου επιχειρήσεων, υπηρεσιών, που θα συγκεντρώνει τους πόρους και τα μέσα για τις μη στρατιωτικές επιχειρήσεις. Και σας καλώ από τη συνάλλευση της Υποεπιτροπής, ε, αλλά και γενικότερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να δούμε αυτό το πολύ σημαντικό ζήτημα, Γιατί οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπόκεινται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο και επαναρχόμενος στη στρατηγική αυτονομία. Νομίζω ότι είναι πολύ περίεργο, να μην πω κάτι άλλο, το εξή. Λαμβάνοντα υπόψη ότι γίνεται στην Ανατολική Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να αγοράζει εξοπλισμό από τη Ρωσία. Θέλουμε στρατηγική αυτονομία για την Ένωση, παραλαμβάνω. Βλέπω όμως κυρίες και κύριοι μια νέα αρχή, ένα νέο ξεκίνημα για την ΚΠΑ, για να πετύχει βήμα-βήμα τη στρατηγική αυτή αυτονομία. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Arnold. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ντανζάν και τελειώνει εδώ ο κατάλογος των αμιλητών. Α, όχι, και ο Τζέφρι Βαν Όρντεν και ο Τζέφρι Βαν Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούν ότι το θέμα είναι αποφασιστικό για το μέλλον της ε, ΚΠΑΣΑ. Και το έχουν καταλάβει και οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στη διάσκεψη του Δεκεμβρίου. Άρα και για αυτό το θέμα και για τα υπόλοιπα που είχαν τεθεί τότε δεν, υπήρξε, δεν σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος. Το Δεκέμβριο το 2013 εννοώ. Ε, πάνω από ένας χρόνος πέρασε και δεν έγινε τίποτα για καλύτερη ή περισσότερη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων της ΚΠΑΣΑ. Απ' την άλλη, από τη μία οι πολιτικές επιχειρήσεις, τα είπε ο Κριστιαν, το πρόβλημά τους δεν είναι το ύψος του προϋπολογισμού των... Εδώ μπορούν να βολευτούν τα πράγματα. Και χρηματοδοτήθηκαν επαρκώς όλες οι επιχειρήσεις. Η λειτουργία τους, η χρήση του προϋπολογισμού αυτού είναι πρόβλημα. Με όλες τις λειτουργίες που σημειώθηκαν εδώ και 15 χρόνια. Σημειώνω αυτά που είπε πανυπροηγούμενοι εμπειρογνώμονες αλλά οι διαπιστώσεις πολλές φορές είναι απλά εμπειρικές. Και αυτό είναι άδικο και για το προσωπικό που χρησιμοποιείται επί τόπου και για την Ευρωπαϊκή Ένωση πολιτικά, διότι διότι η αξιοπιστία της μειώνεται. Μετά υπάρχει το στρατιωτικό πρόβλημα. Έξι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουμε αυτή τη στιγμή. Εκτός από το Μαλί, που, όπου συνεισφέρουν 23 κράτη, οι υπόλοιπες πέντε χρηματοδοτούνται από 5-6 ποτοπολί κρατη κράτη-μέλη. Και τρίτες χώρες είναι αυτές που συμπληρώνουν Τουρκία, Γεωργία και άλλες. για να εφαρμοστεί ευρωπαϊκή στρατιωτική επιχείρηση. Σο, πολύ σοβαρό είναι αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή και η Αταλάντη που θεωρήθηκε μεγάλη επιτυχία μόνο 5-6 χώρες τη χρηματοδότησαν. Είναι λοιπόν σοβαρό το πρόβλημα και άρα η χρηματοδότηση δεν είναι μόνο ότι πάντα οι ίδιοι την κάνουν, είναι και ότι δεν συνεισφέρουν χώρες που θα ήθελαν αλλά που σε περίοδο κρίσης δεν έχουν τα μέσα να το πράξουν. Υπάρχει λοιπόν ένα ζωτικό πρόβλημα εδώ και νομίζω ότι η μόνη λύση, το είπαν και οι συνάδελφοι του ΕΛΚ, είναι η διεύρυνση της Αθηνάς. Ξέρουμε ότι είναι πολύ ακριβές οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και ιδίως η μεταφορά και αυτά δεν τα καλύπτει η Αθηνά. Και αυτό είναι εκείνο που εμποδίζει ορισμένε χώρε μέλη να συνεισφέρουν. Αν δεν διευρυνθεί η Αθηνά λοιπόν, δεν θα γίνει τίποτα, να μην έχουμε αυταπάτε. Και για να τελειώνω, ο δημοκρατικός έλεγχο, κοινοβουλευτικό έλεγχο, και εγώ κοινοβουλευτικό είμαι, θα ήθελα πολύ να μπορώ να πω ότι υπάρχει κοινοβουλευτικός έλεγχος των επιχειρήσεων αυτών, αλλά εδώ ειλικρινά για να τα πούμε, Καμιά φορά κάνουμε επισκέψεις και παρακολουθούμε τη λειτουργία, αλλά οι εκθέσεις μας μετά από τις εκθέσεις, οι εκθέσεις μας μετά από τις αποστολές αυτές έχουν καμία επίπτωση στη λειτουργία της επιχείρησης. Πραγματικά θα ήθελα να μπορούσα να σας πω ναι, ελπίζω να υπάρχει ένα ελάχιστο, μια ελάχιστη επίπτωση, αλλά αν κρίνω από το τι λέει η Κομισιόν και η εξωτερική Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, κάνουν ό,τι θέλουν και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος, επιτρέψτε μου να σας πω ότι μπορεί να μας αρέσει ως ιδέα και έννοια, αλλά δεν λειτουργεί καθόλου πολιτικά. Και αυτό δεν το λέω για την αναθεώρηση των χρηματοδοτήσεων. Και τέλος, το άρθρο 44, η μόνιμη δομημένη συνεργασία, αυτό είναι πρόβλημα που θα μπορούσε να λύσει, να διορθώσει τα πράγματα, αλλά ξέρουμε τι γίνεται από τις κυβερνήσεις. Το κλειδί είναι στις πρωτεύουσες των χωρών μελών και ξέρουμε ότι πολλές από αυτές δεν θέλουν να παίξουν το παιχνίδι. Και αυτό μειώνει πολύ το τι μπορούμε να κάνουμε. Πρέπει να το γνωρίζουμε δεν λέω να μην κάνουμε συστάσεις, αλλά να ξέρουμε ποια είναι τα όρια που θα αντιμετωπίσουμε μπροστά μας από τις κυβερνήσεις. Χριστό. Τζέφρι Βαν Όρντεν, συντονιστής των συντηρητικών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακούγοντας τη συζήτηση αυτή διαπιστώνω ότι υπάρχει εδώ κάποια έλλειψη εντιμότητος, ειλικρινίας. Δεν αναγνωρίζεται δηλαδή η αχρηστία της ΚΠΑΣΑ. Δεν παίζει κανένα ρόλο, δεν θα είχε καμία διαφορά άμα δεν υπήρχε καμία αποστολή της ΚΠΑΣΑ. Ούτε για την ασφάλειά μας, ούτε για την ασφάλεια των χωρών που υποτίθεται ότι ωφελούνται γενικότερα. Ποιος είναι ο ρόλος που θέλουμε να παίξουμε. Να δημιουργηθεί λέει στρατηγική αυτονομία της Ένωσης ή να αυξηθεί η ορατότητά της διεθνώς. Όλα δηλαδή είναι θέμα θεάτρου. Ότι τάχα έχουμε κάποιο ρόλο να παίξουμε διεθνώς και ελέγχουμε δυνάμεις κλπ. Βέβαια αν θέλουμε να μειώσουμε τη διαφορά μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών αποστολών, θα έπρεπε να πούμε ότι αν βγάλουμε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν γίνεται τίποτε άλλο δεν γίνεται από την ΚΠΑΣΑ. Άρα η όλη συζήτηση είναι φαντασιώδης. Και αυτό είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους και οι πολίτες της χώρας μας σηκώνουν ψηλά τα χέρια και λένε μα κοίτα τι γίνεται στην Ένωση. Τίποτα δεν γίνεται. Και όλα αυτά που λέμε σήμερα είναι εκτός πραγματικότητας και δεν χρειάζονται. Τα κράτη-μέλη γνωρίζουν πλήρως τι πρέπει να κάνουν με τις δικές τους δυνάμεις και μερικές από αυτές μιλάνε σοβαρά για στρατιωτικές επιχειρήσεις και παίζουν πραγματικό ρόλο, αν χρειάζονται λοιπόν στρατιωτικές επιχειρήσεις διεθνώς, υπάρχουν δομές και οργανώσεις που το συντονίζουν. Υπάρχει το ΝΑΤΟ και υπάρχουν και άλλες εθελοντικές συμμαχίες. Το τελευταίο που θα χρειαζόμασταν θα ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση να εφεύρει έναν ακόμη ρόλο για τον εαυτό της. Είναι γελίο. Thank you. Um, now, uh, Τώρα θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Επιτρέψατε μου όμως να σας δώσω κάποιες πληροφορίες. as he was mentioned by... Να δούμε ποιοι θα πούν κάποιες καταληκτικές παρατηρήσεις. Επειδή ο κύριος Γκάλερ ε, αναφέρθηκε ονομαστικά από δύο, αν θυμάμαι καλά, συναδέλφους θα πάρει το λόγο, έπειτα ο καθηγητής Τέρπα, οι δύο εισηγητές, πιστεύω ότι θα πρέπει να απαντήσουν τις ερωτήσεις η κύριη Κουκαντάρπαν και ίσως και η κύριη Ντίν και Μίλλερ. Κύριε Γκάλερ, εσύ σύντομα. Κοιτάξτε, να αντιδράσω επειδή τέτοιο θέμα. Συνάδελφε, ε, μάλλον με παρεξηγήσετε, εγώ δεν εννοούσα ότι όλα τα κράτη θα πρέπει να συμμετέχουν σε όλες τις επιχειρήσεις με τις δικές τους δυνάμεις. Δεν πρόκειται περί αυτού. Εγώ θέλω να πω ότι επειδή όλοι αποφασίσαμε ομόφωνα ότι κάτι πρέπει να κάνουμε, ο καθένας ανάλογα με τη συμμετοχή του στον προϋπολογισμό θα πρέπει να συμμετέχει και στο μηχανισμό Αθηνά και να δούμε ε, ποιος το κάνει καλύτερα. Και με αυτόν τον τρόπο, κατά την άποψή μου, ε, θα προκύψει ένας ε, μηχανισμό μηχανισμός ε, που θα ε, προσφέρει και το ποσοστό το οποίο θα προσφέρει όλος ο μηχανισμός θα αφαιρείται από το σύνολο του προβλογισμού. Αν είναι 8% το υπόλοιπο 92% θα καλύπτεται από τον προπλογισμό. Θα υπάρχει δηλαδή ένας στρατός, αν θέλετε, οι δυνάμεις που δεν θα καλύπτονται πλήρως από τον ε, προϋπολογισμό. Το άλλο, το στρατιωτικό και μη μη στρατιωτικό, βεβαίως και είναι σημαντικό στην κεντρική αφρικανική δημοκρατία. Εκεί λέμε ότι θέλουμε να επιτύχουμε ε, μια αλλαγή, μια μεταρρύθμιση στην, ε, στις αστυνομικές δυνάμεις το ε, μη στρατιωτικό σκέλος μπορεί να χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ξεχωριστά τώρα τι θα γίνει τα αεροπλάνα θα μπορούν να πετάνε στο πλαίσιο μιας επιχείρησης που αυτοί θα μεταφέρουν τους ε, εκπαιδευτές. Δηλαδή αυτή, αυτός ο διαχωρισμός ε, πολλές φορές είναι τεχνητός και εγώ απλά ήθελα να πω ότι πρέπει να είμαστε πιο ρεαλιστές. Ο καθηγητής παρακαλώ πολύ σύντομα. Ναι, πολύ σύντομα. Επανέρχομαι σε δύο-τρία στοιχεία. Καταρχάς, ότι δηλαδή πρέπει να έχουμε υπόψη μας τι προβλέπεται από τις συνθήκες και μέσα σε αυτό το πλαίσιο να κινούμαστε η εξέλιξη των συνθήκων και εδώ βλέπω και το ρόλο του Κοινοβουλίου. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερο, δύο επίπεδα υπάρχουν, το τεχνικό και το πολιτικό. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές λύσεις που φαίνονται γρήγορα υλοποιήσιμες, εφικτές, το Shared Service Center, από την τεχνική πλευρά, αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα που άπτονται καθαρά του πολιτικού επίπεδου και εδώ. Είναι επίσης ρόλος για το Κοινοβούλιο να τοποθετηθεί και στα δύο επίπεδα. Τέλος, κυριαρχία ε, όσον αφορά τον προϋπολογισμό, στρατηγική αυτονομία, νομίζω όλοι συμφωνούμε με τον κοινό αυτό στόχο. Τα κράτη-μέλη σίγουρα μπορούν να, να συμμετάσχουν ή να μην συμμετάσχουν γιατί έχουν ε, την εθνική κυριαρχία σε ό,τι αφορά την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Να έχουμε συμμετοχή αλλά κάρτ σε όλους τους τομείς δεν θα λειτουργούσε αυτό. Δεν ξέρω. Για το συγκεκριμένο τομέα θα μπορούσε ίσω, αλλά για φανταστείτε να εφαρμοστεί το ίδιο σε όλους του τομεί δραστηριότητα τη Ένωση. δεν θα λειτουργεί πλέον η Ένωση. Η πρόεδρο, σας ευχαριστώ κύριο Κούκαν. Ευχαριστώ κυρία πρόεδρε, πάρα πολύ σύντομα. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχά όλου του συναδέλφου αλλά και τους προσκεκλημένου που συμμετείχα στη συζήτηση αυτή. Σας ευχαριστώ για τις απόψεις τους, γιατί είναι καλό να πιάσουμε το σφιγμό, να ξέρουμε τι πιστεύει ο καθένας. Ευχαριστώ τον καθηγητή Τέρπαν και τους κυρίως από την Κομισιόν και την ΕΙΕΔ που έδειξαν και την ε, τιμότητά τους ε, να συνεισφέρουν. Σε ό,τι αφορά τις δύο ερωτήσεις του συναδέλφου από την Άλντε, δεν μπορώ να δώσω πλήρη απάντηση, αλλά μπορώ να του πω ότι θα τις λάβω τις ερωτήσεις του υπόψη όταν θα περάσω στη σύνταξη της έκθεσης αν μπορώ να καταλήξω σε κάποιο συμπέρασμα από την όλη συζήτηση, μπορώ να πω ότι στην έκθεσή μου θα προσπαθήσω την, ε, τον οικονομικό έλεγχο και την εποπτεία του Κοινοβουλίου να τον αυξήσω, θα στηρίξω την αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών και θα ζητήσω ξεχωριστά κονδύλια στον προϋπολογισμό για την κάθε επιχείρηση αποστολή και φιλοδοξώ να συντάξω μια έκθεση που θα μπορεί να επηρεάσει πραγματικά τη μελλοντική ΚΕΠΑ, η ΚΠΑ. Και να είναι μια πραγματικότητα και όχι ουτοπία. Ευχαριστώ. Και uh, oh, ο Mr. Indrek Ο α, απουσιάζει. Ο πρόεδρος Αχτουή θα ήθελε μήπως να πει κάποια καταληκτικά σχόλια. Το συμπέρασμα είναι προφανώς προσωρινό, αλλά με ενδιέφεραν πάρα πολύ όσα άκουσα, ιδίω τον καθηγητή Τερπάν και τους υπόλοιπους και νομίζω ότι καλή ιδέα είναι να έχουμε αναλάβει αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας για την πάσα από κοινού οι δύο επιτροπές. Ο προϋπολογισμός τελικά είναι καθρέφτης καθρέφτης των μέσων που διαθέτουμε και από αυτή την άποψη δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτας. Παρά το ότι πρόκειται για πολιτικές αποστολές 300 περίπου εκατομμυρίων θα χρειαστεί να πληρώσουμε. Όταν μιλάμε για την ανάγκη γρήγορης παρέμβασης πρέπει να έχουμε τα μέσα να το πράξουμε και αυτό αφορά κυρίως την αξιοπιστία μας ο προπολογισμό βέβαια προκύπτει αποκλειστικά από τα κράτη-μέλη αφού δεν έχουμε πια ιδίους πόρους. Άρα ο προϋπολογισμός εξαρτάται από τα κράτη-μέλη. Και αυτό δυσκολεύει πολύ τα πράγματα. Φυσικά πρέπει να σεβαστούμε τις συνθήκες, αλλά μου φαίνεται ότι ο λόγος ύπαρξής μας εδώ είναι και η άσκηση πολιτικής. Και το θέμα είναι αν η Ευρώπη μπορεί και πρέπει να έχει δικαιοδοσίες σε θέματα ασφαλείας και άμυνας ή όχι. Από το 1954 ζητήθηκε η δημιουργία μιας κοινή πολιτικής άμυνας, αλλά αρνήθηκαν τότε τα κράτη-μέλη. Τώρα όμως που έχουμε την παγκοσμιοποίηση, τι μπορούμε να πούμε στους συμπολίτε μας. Βλέπω κι εγώ τι ζητάμε εδώ και τι συζητάμε. Όταν επιστρέφω όμως ενώπιον των συμπολιτών μου και των εκλογέων μου, δεν μπορώ να τους τα εξηγήσω πώς μπορεί ο πολίτης να είναι αλληλέγγυος με την Ευρώπη για θέματα ασφαλείας και άμυνας. Ζούμε σε μια φαντασίωση όπως είπε κάποιος ή στην πραγματικότητα. Έχουμε πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο που μας δεσμεύει από το 14 στο 20 αλλά υπάρχει και μια ρήτρα αναθεώρησης και θα ήθελα η έκθεση αυτή πρωτοβουλίας να μαζέψει επιχειρήματα για μια πιθανή αναθεώρηση του προϋπολογισμού μας. Ήδη προετοιμάζουμε τον προϋπολογισμό του 16 και δεν αφιβάλλω ότι θα ήταν ενδιαφέρον να ακούσουμε τι έχουν να μας πούν οι εισηγητές ως προτάσεις. Σημείωσα πάντως αυτά που είπε ο καθηγητής και βρισκόμαστε στα όρια της φαντασίωσης ή αν όχι των κύριων στοιχείων που θέλουμε να εφαρμοστούν ως ασφάλεια και άμυνα. Και αν δεν υπάρχει κοινή ασφάλεια και άμυνα, πώς να υπάρχει κοινή εξωτερική δράση. Ζούμε λοιπόν μια αποφασιστική φάση στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση και το θέμα είναι αν μπορούμε ή αν πρέπει να κάνουμε αυτό το βήμα. Εγώ είμαι καινούργιος κοινοβουλευτικό, τώρα έμαθα για το μηχανισμό της Αθηνάς είναι περίεργο πράγμα εκτός προϋπολογισμού, είναι αλακάρτης φορές ότι όποιο κράτος θέλει παρέμβαση πρέπει και να την πληρώσει και μετά ζητάει την άδεια από τους εταίρους του κτλ. αυτές τέτοιου είδους μηχανισμοί δεν μπορούν να επιβιώσουν. Ευχαριστούμε κύριε μου. θα αποφασιστούν όλα αυτά από την Επιτροπή Προπολογισμών στις 26 Φεβρουαρίου μετά η διορία κατάθεση τροπολογιών λίγη στις 3 Μαρτίου το μεσημέρι και εδώ τελειώνει η κοινή συνεδρίαση προϋπολογισμών και υποεπιτροπής ασφαλείας και άμυνας. Ευχαριστώ. Δεκάλεπτο διάλειμμα και μετά η κανονική μας συνεδρίαση. Ευχαριστώ. <laughs>